Euh, Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Με συγχωρείτε που ξεκινάμε με καθυστέρηση της εργασίας. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι χθε συμπεριλάβαμε δύο τροποποίησεις στην ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, το σημείο 11, το οποίο αφορά την εξέταση των τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Μάκιντάιρ, θα εξεταστεί μετά το σημείο, ή μάλλον το σημείο 11 θα εξεταστεί μετά το σημείο 21. Πρόκειται συγκεκριμένα... Α, όχι, δεν είναι σχέδιο γνωμοδότηση, είναι σχέδιο έκθεση. Έκθεση πρωτοβουλίας τη κυρία Μακιντάι. Για τη δημιουργία φιλόξενου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις Δεύτερη τροποποίηση που συμπεριλάβαμε χθε, αναβάλλεται για το τέλος των εργασιών μα, δηλαδή μπαίνει ως τελευταίο σημείο τη μερίσιας διάταξη μετά το σημείο 25, το σημείο 13, το οποίο προβλεπόταν να εξεταστεί χθε και αφορά ανταλλαγή απόψεων για τις διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με το Ταμείο για τους Άπορους. Κυρία Έμερ Κοστέλο, η συγγήτρια και την ευχαριστώ που αυτή την αλλαγή. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, ε, έχουμε το σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Το θέμα είναι η κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. Πρόκειται για εκθέση πρωτοβουλία της Επιτροπής μας, με εισηγήτρια την κυρία Βίλια Μπλινκεβιτσιούτε. Έχουμε 144 τροπολογίες, ε, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε και βέβαια έχουν και 27 συμβιβαστικές τροπολογίες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε εισηγήτρια. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που κατέθεσαν τροπολογίες, 144 στον αριθμό, καταφέραμε να συντάξουμε 29 συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες αφορούν όλες τις συντολογικές σκέψεις, τα ρησάιτρας και σχεδόν όλες τις παραγράφεις του κειμένου. Είχαμε μια συνάντηση με τους σκιώδες εισηγητές την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όπου συζητήσαμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. 27 εκ των 29 είχαμε συζητήσει βέβαια τότε και εγώ πρόσθεσα δύο στη δεύτερη έκδοση των συμβαστικών τροπολίων και θα ήθελα να σας τις παρουσιάσω. Η πρώτη νέα συμβαστική αφορά ε, το recital GA λατινικό για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους που το 2012 αντιστοιχούσαν ε, στο 15% της αγοράς εργασίας. Πρόκειται δηλαδή για ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού και συχνά ε, τα άτομα επιλέγουν το καθεστώ του αυτοαπασχολούμενο διότι έτσι ε, δεν εντάσσονται στην κατηγορία των μακροχρονίων ανέργων. Ουσιαστικά έχω ε, συγκεντρώσει σε μία τροπολογία πολλές παρόμοιες τροπολογίες. Δεύτερη νέα συμβιβαστική αφορά το νέο τμήμα 5α που τροποποιεί κατά κάποιο τρόπο τη διατύπωση της προηγούμενης τροπολογίας για τη διατήρηση των ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας που έχουν εμπειρία, έχουν εμπειρία εργασιακή και δεν θα έπρεπε να τα θεωρήσουμε σε καμία περίπτωση οικονομικό ή κοινωνικό βάρος. Τροπολογία τη κυρία Όμεν Ρόιταν, αρχικά τη στηρίζω. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν και με τι δύο νέε αυτέ συμβιβαστικέ τροπολογίε. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι στην συνεδρίαση αυτή των σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε και σχεδόν επί του συνόλου των συμβαστικών τροπολογιών. Κύριο θέμα ήταν ε, η η ανεξαρτησία αυτών των ε, εργαζομένων, τι πρέπει να γίνει για να έχουν την ενημέρωση που πρέπει σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Συμβαστικές τροπολογίες επίσης καθορίζουν τις αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών και πού υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Στην τελευταία συμβαστική πρόταση γίνεται λόγος για τους κοινωνικούς εταίρους. Ελπίζω να γίνει δεκτή. Θα ήθελα να την δεχθούν και οι συνάλφοι του ΕΛΚΑ, που έχουν άλλωστε καταθέσει πολλές τροπολογίες για τους κοινωνικούς εταίρους. Χθε το πρωί στείλαμε τη δεύτερη εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών σε όλους τους και όλες τις ηγητές. Προσπάθησα να συμπεριλάβω σε αυτές όλες τις ε, προτάσεις που είχαμε συζητήσει μέχρι τώρα. Περιμένω τώρα λοιπόν να ακούσω τα σχόλια, τις απόψεις ε, των σκιωδών εισηγητών. Ελπίζω να έχω ολοκληρώσει μέσα στη βδομάδα, ώστε να μπορέσουμε στις 5 Δεκεμβρίου την επόμενη εβδομάδα να ψηφίσουμε. Αυτά είχα να πω. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας, τις υποδείξεις σας. Ποιοι είναι οι συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρεύουν, Φιλμπενιό. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν καταφέρα να παρευρίσκομαι στη συνάντηση σχεδόν την περασμένη εβδομάδα. Είχα τρία ραντεβού. Θα ήθελα να σχολιάσω τις συμβιβαστικές εδώ. Θα στείλω τα σχολιά μου και γραπτός. Αργότερα. Υπέβαλα αρκετές τροπολογίες. Οι περισσότερες έγιναν δεκτές από την εισηγήτρια. Πιστεύω είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αρμοδιότητα κρατών μελών, αλλά σε κάποιο βαθμό μπορεί να συντονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε διάφορες δηλώσεις για τα ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των διαφορών κρατών μελών. Χαίρομαι λοιπόν με τις διατυπώσεις της συμβαστικής C&D. Στη συμβαστική D δεν συμφωνώ με τη διατύπωση στο τελευταίο τμήμα. Θα ήθελα οι λέξεις widely και glaring να καταργηθούν και το leading να αλλάξει σε could lead στη συμβιβαστική F. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που έλαβε υπόψη την τροπολογία μου του could be useful. Εκπροσωπεί την ε, ψευδής ε, περίπτωση αυτοαπασχόλησης. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες. Χαιρόμαι τις τροποποίησεις του Αλαντέμου βάσει των σχολείων της τελευταίας συνάντησης σχεδόν. Η συμβαστική ΕΝ επίσης είναι πολύ ικανοποιητική. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε όλους τους δικαιούχους που παραμένουν ε, με τη βούλησή τους στην αγορά εργασία και ειδικότερα όσον αφορά τη μεταφορά ικανοτήτων. θα προτιμούσα να λέμε guaranteed access αντί για guarantee, γιατί η κοινωνική ασφάλιση στα περισσότερα κράτη-μέλη βασίζεται στο καθεστώ του ενδιαφερομένου και μπορεί να βασίζεται σε προποθέσει. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τι αρμοδιότητε των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Στη συμβαστική P unjustified της μέσω πρέπει να είναι η σωστή διατύπωση για, τις περιόδους, για το κομμάτι που αφορά της εγγύους. Αλλιώς μένουμε σε μια κατάσταση όπου μια εγγύους γυναίκα δεν θα μπορούσε να απολυθεί για ε, κακή συμπεριφορά, το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε εδώ. Θα στείλω τα υπόλοιπα μου σχόλια, γραπτό παρόλα αυτά. Δεχόμαστε τι περισσότερε συμβιβαστικέ. Ε, Όπω βλέπετε, είναι πολύ συγκεκριμένα, αφορούν λεπτομέρειε στα σχόλια μου. Ε, γενικότερα, με το γενικό τρόπο συμφωνούμε. Ε, Ευχαριστούμε. Κύριος Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ είμαι ικανοποιημένο ε, που έχουμε αυτή την έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Όταν μιλάμε για κοινωνική προστασία στην Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει αρμοδιότητα κρατών μελών, αλλά φυσικά μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, για κάποιου στόχου σε θελοντική βάση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που βρισκόμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα και που καταλήξαμε σε κάποιου συμβασμού. Στι περισσότερε περιπτώσει είμαι βέβαιο ότι παραμένουν κάποια εκκρεμή ζητήματα, αλλά είμαι σίγουρο ότι μέχρι τις, 5, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θα καταφέρουμε να καταλήξουμε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε, θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, εν συντομία να ευχαριστήσω τον κύριο Μπένιον, να ευχαριστώ και τον κύριο Σαββασοντόρ για την ε, συνεργασία μας οι παρατηρήσεις του κ. Μπενίων ελπίζω να μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν με σίγουρη στη συνέχιση των εργασιών μας. Τον ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρος. Δεδομένων αυτών λοιπόν θα ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου. Οι φιλελεύθεροι έχουν ακόμα να κάνουν κάποιες προσαρμογές αλλά ελπίζω να μην θέσουν σε κινδυνό τις συνθήκες προστασίας που προτείνονται ειδικότερα για τις εγγύους. Καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά τώρα έχουμε κερδίσει. καλύψει το χρόνο που χάσαμε. Συμφωνούν οι ομάδες να εξετάσουμε το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλαδή να κάνουμε τον απολογισμό των διαπραγματεύσεων feed του Ταμείου για την Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς Όχι, δεν συμφωνεί ο κύριος Σέρκας για τους σοσιαλιστές, δεν συμφωνεί. Δεν μπορούμε λοιπόν Αφού έχουμε τα πράγματα να περάσουμε στα διάφορα τότε ίσως τώρα. Στα διάφορα ήθελα απλά να σας αναφέρω την εξέλιξη των συζητήσεών μας για τα θέματα που ανέφερα χθες για τα διάφορα σε σχέση με τις εργασίες των συντανιστών όταν συναντήθηκαν με τον Επίτροπο Αντόρ για την υλοποίηση των συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Όπω ανέφερα χθε, 9 Οκτωβρίου συναντήθηκαν οι συντονιστέ και κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση συμφώνησαν όλοι για ανταλλαγή απόψεων με τον Επιτροπό Αντόρ για το θέμα τη υλοποίηση των συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Επίσης, συμφώνησαν να δημοσιεύσουν ένα δελτίο τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Το δελτίο αυτό τύπου κυκλοφόρησε τέλος περασμένης εβδομάδας την Παρασκευή μετά από τη συνάντησή τους που έλαβε χώρα την Πέμπτη πρωί. Κάποιες ομάδες ε, μου είπαν, με ενημέρωσαν ότι δυσκολεύονταν να υποστηρίξουν το δελτίο τύπου όσο έχει Σήμερα λοιπόν το πρωί θα κυκλοφορήσει, θα δημοσιευτεί ο απολογισμός των εργασιών έτσι όπως εξελίχθηκαν με το δικό μου όνομα. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κανένα τηλεφώνημα, έχετε 5 λεπτά, διότι θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες τις 9 και μισή, ζητώ συγγνώμη από τους δίρμηνες που δεν θα κάνουν τίποτα για 5 λεπτά, αλλά σας το υπόσχομαι Θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε ώστε να προχωρήσουμε στις ψηφοφοριες Έχουν όλοι οι συνάδελφοι τις κάρτες ψηφοφορίας τους. c'est le cas, nous allons tout d'abord au point. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 15 να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για την 7η και 8η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περίοδου 2007-2013. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, του συναδέλφου Αντάμ Κόσο. Για την παράγραφο 1 έχουμε την τροπολογία 1. της Μαριάν Χάρκεν με μια επιπλέον ε, διόρθωση ορθογραφικού λάθους ε, είναι υπέρ, ο εισηγητής ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην παραγραφή 1 τροπολογία της Elizabeth Schroeder είναι υπέρ, ο εισηγητής υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρία αντιγόνες Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1 τροπολογία 4 ιδίας ε, με προφορική τροποποίηση τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροπολογία στην παραγραφό 2 συμβαστική α από τέσσερις ομάδες με προφορική τροπολογία ε, υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία όχι ψηφίζουμε λοιπόν όλη τη συμβαστική α υπερκατά αποχές εγκρίνεται στην παράγραφο 2 τροπολογία 9 Αντιγονής Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της Ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβιβαστική β 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 ε, τροπολογία 13 Αντιγονής Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 D από δύο ομάδες υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Παραγωγή 4. Συμβαστική C τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγωγή 4. Τροπολογία 18. Αντίγονη Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το κείμενο ηλεκτρονικά. Έρχεται ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ψήφισαν πέρα πέρας ψηφοφορία. 30 υπέρ, ε, μία ψηφο κατά, καμία αποχή, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, Περνάμε τώρα στο σημείο 16. Θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλία για τι ε, αποτελεσματικέ επιθεωρήσει εργασία ω στρατηγική για την βελτίωση των συνδικών εργασία στην Ευρώπη έκθεση της συναδέλφου Γιούτας Στάινροκ. Στην παράγραφο 1 ψηφίζουμε τη συμβαστική σε από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα στην παράγραφο 1 υπάρχει συμβαστική CA. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 45 του κ. Πουπάκη, όπου έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το σύνολο της τροπολογίας χωρίς τις λέξεις αναδιοργάνωση είτε. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης αυτών των δύο λέξεων. Ε, αναδιοργάνωση είτε. Υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 46, η Καριμάντελη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 2, συμβαστική ιδέα από τέσσερι ομάδε υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 51 του κυρίου Πουπάκη, δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα Χωρί τι λέξει που προκύπτουν εν μέρη, ε, ε, έως και σχέση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική ε 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα για την παράγραφο. Συμβαστική εα από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 55 μπουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 πουπά... πουπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 αντελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 ντελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. 59 Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4. Τροπολογία 60 Ιούτα Στάινρουπ. Με προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 4 πάντα τροπολογία 61 τη συζήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 της συζήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφό 5 τροπολογία 63 εσαϊά είναι τροπολογία απάλυψης, άρα όλοι όσοι ε, είναι υπέρ τη ΕΦ δεν μπορούν να την ψηφίσουν. Ψηφίζουμε την 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστικής F τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε είμαστε στην παράγραφο 6, ίδια κατάσταση. Τροπολογία πάλιψη, 70 της κυρίας ε, του Εσαϊά. Ποιοι είναι υπέρ του 70. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 80, Κρίστενσεν, υπέρ. Κατά αποχές. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την 80. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 16 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8 συμβαστική H. Τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 συμβαστική I. Τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη συμβαστική I. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 22 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 93 της συγκήτριας υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 94, που πάει και υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Συμβαστική J από τρεις ομάδες υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 99 της συγκήτριας υπέρ, κατά Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την 99. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 16 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. 100 της συγκήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Τρεις τροπολογίες απάλληψης που δεν θα μα επέτρεπε να ψηφίσουμε τη συμβαστική ΚΑΠΑ. Οι τροπολογίε 101-103 να τι ψηφίσουμε από κοινού υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική ΚΑΠΑ από τρει ομάδε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά την παραγράφο 11 τροπολογία 106 Λαντοβέτσικα και άλλων υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 12 συμβαστική L από τρει ομάδε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάντα για την παράγραφο 12 η τροπολογία 109 Χέντελ είναι συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική SA από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12 τροπολογία 113 Κρίστενσεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 Ντελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Συμβαστική μη από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13. Συμβαστική νη από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Τροπολογία απάλληψη που δεν θα σε επέτρεπε να ψηφίσουμε την ε, συμβαστική όμικρο. Ποιοι είναι υπέρ τη 118 του ΜΠΑΚ. Υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Συμβαστική όμικρο από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε. Α, καλά. Να ελέγξουμε τη συμβαστική όμικρο να έρχεται. Ένας ε, σοσιαλιστής παραπάνω. Α, ωραία. Ωραία. Έφυγε. Πέρασε. 22 υπέρ, 13 κατά. Σαφή έγκριση. 122 Handel είναι συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 14 τροπολογία 124 τη ηγήτριας υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 15. Συμβαστική ΠΕ από τρει ομάδε υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 16. Συμβαστική Q από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Ίδια κατάσταση συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 17 τροπολογία 140 Λούντιξον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 μπαχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 17α νέα παράγραφος μετά τη 17 έχουμε την τροπολογία S από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 18 συμβαστική τάφα από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 19 Τροπολογία πάλιψης. Εσαγιά. 150 που σήμερα δεν θα ψηφίζαμε τη συμβαστική γιου από τρεις ομάδες. Υπέρ. 150. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική γιου από τρεις ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 19 η τροπολογία 160 καταπίπτει, οπότε είμαστε στην παράγραφο 20, τροπο, συμβαστική Β από τρεις ομάδε υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 21, 166, για και Σκριτλεύσκα, που θα κατέριπτε τη συμβαστική W. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 166, υπέρ, λοιπόν κατά απόχέ απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική W από τέσσερι ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Τροπολογία 171. Ντελή έχει αποσυρθεί. Αλλά έχουμε την τροπολογία 172. Σλοβιέτσκα και Σκριντλεύσκα που θέλει να απαλείψει. Οπότε θα καταρριπτόταν η συμβαστική χ. Ποιοι είναι υπέρ της 172. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική χ από τρεις ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Y στην 23. Από τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 23, τροπολογία 182, μπουλό, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24, συμβαστική Z από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 24, έχουμε τη συμβαστική ΑΑ από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφή 24, τροπολογία 188, Στάινρουκ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα μετά την παράγραφη 24, τροπολογία 189, Ντελή, υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγξουμε την 189. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 21 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 25 έχουμε τρεις τροπολογίες απάλληψης. 190 έως 92. Οπότε θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αν εγκρίνονταν τη συμβαστική ΒΒ που έχουν ε, υποβάλει το ΕΛ, οι σοσιαλιστές, ε, φιλελεύθεροι και πράσινοι. Ποιοι είναι υπέρ της απάλληψης κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική ΒΒ από τέσσερις ομάδες ε, που τις προανέφερε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Τρεις ε, τροπολογίες απάλληψης 196 έως 198 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε λοιπόν την συμβαστική CC τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 26, τροπολογία 202, δελή, υπέρ. Υπέρ έλεγα. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγράφος 27. Δύο απαλληπτικές. 203 Εσαγιά και 204 Ορί. Οπότε θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την ΤΕΝΤΕ. Ποιοι είναι υπέρ της απάλληψης. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική ΝΤΕΝΤΕ από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το παράγραφο 27, τροπολογία 209 Χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 28. Τέσσερις τροπολογίες απάλληψης. 210 έως 213. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική ε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29. Πέντε τροπολογίες απάλληψης. 216 έως 220. Εσάγια Μπέκερ, Μπαχ, Ορί, Γιασλοβιέτσκα και Σκριτσλεύσκα. Ίσως είναι ΠΠΕ, ε, ίσως είναι έλκολοι αυτοί. Ποιοι είναι υπέρ της απάλληψης 29. Κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την απάλληψη της παραγράφου 29. Ψήφισαν όλοι πέρας. 19 υπέρ, 17 κατά. Η παράγραφος 29 απαλήφεται. Ο, περνάμε τώρα ε, στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 που προτείνει, όχι, στις αιτιολογικές αναφορές που θέλει μια νέα μετά 33. Χέντελ 1 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, συμβαστική α, από τέσσερις ομάδες. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ιδεολογική σκέψη α, τροπολογία 6, μπενιού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάντα μετά την ιδεολογική σκέψη α, η τροπολογία 7, του ιδίου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, ντελή, υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τροπολογία 8 της ε, Ντελή η υπέρ. Ε, πάλι ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Πέρας. 28 υπέρ. 6 κατά. Δεν χρειαζόταν και τόσο πολύ. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 9 Χέντελ υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 9. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 15 υπέρ, 16 κατά. Απορρίπτεται. Αλλά έπρεπε να ελέγξουμε. Τροπολογία 10 μπουλόν υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 11 χέντελ υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 12 μπουλόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη Β η 14 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί είναι γλωσσικό θέμα ψηφίζουμε τη 15 Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την αιτιολογική σκέψη Β 16 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 Ντελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 Τη συγκίτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σε συμβαστική β από 4 σώματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη d τροπολογία 22 για Σλοβιέτσκα Σκριντλεύσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την αιτιολογική σκέψη Δ, τροπολογία 23, ε, υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 23. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 19 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή. 23 εγκρίνεται. Πάντα μετά την τολογική δέλτα, 24 λέγνερ υπέρ, κατά αποχές. Ε, υπέρ ξανά, υπέρ παραγωγή 24. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 24. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 16 υπέρ, 16 κατά, 4 αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25, Στάνιο υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, Α, να ελέγξουμε την 25. Καλά, να ελέγξουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, 28 κατά, λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, έλεγα 27 υπέρ, 8 κατά. Κάτι έγινε γιατί τώρα περνάει, περνάει πάρα πολύ καθαρά. Κάτι έγινε στη μυστική ψηφοφορία μετά την τολική ε, τροπολογία 26 του κ. Πουπάκη με προφορική τροπολογία όπου δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία. Ψηφίζουμε την 26 όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 26. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 16 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 Κοστέλο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Ντελή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 Ισηγήτρες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 του κυρίου Ποπάκη με προφορική τροπολογία για την οποία υπάρχει αντίθεση. Η 30 τροποποιηθήσα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 Ντελή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 της ηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 η ηγήτρες υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 33 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας 16-16-4 απορρίπτεται 34 της ηγήτρες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 της ηγήτρες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 της ηγήτριας με προφορική τροπολογία π.χ. είναι υπέρ 36 όπως έχει τροποποιηθεί κατά αποχές εγκρίνεται 37 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 Τη ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονικά άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας 22 υπέρ 13 κατά 0 αποχές συγχαίρουμε την εισηγήτριά μας οι οποίοι είναι πολύ ικανοποιημένοι. Περνάμε στο σημείο 17 της μερίσιας διάταξης. Έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γυναικών. μετανάστρες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ψηφίζουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, όπως ε, την συνέταξε ο Μάρτιν Κάστλερ. Στην παράγραφο 1, συμβαστική α από τέσσερι πολιτικέ ομάδε υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, συμβαστική β από τέσσερι ομάδε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 1, τροπολογία 7, μια κονσάρι υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 8 τη ιδέα υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της Ιδίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραφορή συμβαστική C από τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, το 16, της Λίσσα για κονσάρι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17, Γιουτα Στάνρουκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 18 για κονσάρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 3 έχουμε τη συμβαστική δέλτα από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3 τροπολογία 22 κάστλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 Στάινουρκ υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, 16 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24, Κλοντέτ Μπαλτατσίνο. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται στην πάραφο 4, συμβαστική ε, από... Από τι θέλετε, Ελιζαμπέτ Σρέντερ, για την ε, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ως πράσινοι είμαστε κατά της προφορικής τροπολογίας. Τρία άτομα πρέπει να αντιτίθενται στην προφορική τροπολογία για να καταπέσει. Από ό,τι φαίνεται με τις παρεμβάσεις του κοινού όμως, που αυτό δεν επιτρέπεται. Για να δούμε. Ωραία. Ε, δεν γίνεται δεκτή προφορική τροπολογία. Υπάρχει επαρκή αριθμό διαφωνούντων, άρα ψηφίζουμε χωρίς την προφορική τροπολογία την ε, που εκπροσωπούνται σε αυτήν τρει ομάδε παρόλα αυτά. Υπέρ τη συμβαστική ε. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική ε. Παράγραφος 5, τροπολογία 28, Μάρτιν Κάστλερ, ε, υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 για κονσάρι είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε τροπολογία 29 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα, ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 4 αποχές. Η τροπολογία 29 απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 5, συμβαστική F από 4 πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 31, Αντιγόνης Παπαδοπούλου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 32, Γιούτα Στάινρουκ υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε την 32. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 16 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 4 αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 Στάνιρουκ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 Νάντια Χίρς υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα περνάμε στο σημείο 19. Σχέδιο έκθεσης. όνομά μου. Τροποποίηση της οδηγίας 2010 κάθετος 17 του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής καθεστώτος της Μαγιότ. Ως εισηγήτρια θέλω να σας πω ότι τη 2 και την 5 τροπολογίες τις έχω αποσύρει. Ε, σε ό,τι τον τίτλο Solemn Form, το άρθρο 2, το άρθρο 4, έχω τέσσερις τροπολογίες, 1, 6, 8 και 9 συγκεκριμένα, ταυτόσιμες, με κοινό στόχο. Θα σας πρότεινα λοιπόν να τις ψηφίσουμε από κοινού. Δεν ακούτε τη μετάφραση? Τι συμβαίνει? Is it becoming better and better again? Βελτιώθηκε η κατάσταση? Βελτιώθηκε η κατάσταση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 1, 6, 8, 9, τις τέσσερις από κοινού, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Στο άρθρο 1, τροπολογία 13, Σρέντερ. Διαγραφή. Είναι κατά η συγκεκριά υποφαινομένη, δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην αιτιολογική αναφορά έχει αποσυρθεί 2, άρα ψηφίζουμε την 10, πατρίς στη ρολιά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην αιτιολογική αναφορά 5, έχουμε το 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στις αιτιολογικές σκέψεις τώρα, στην 1, έχουμε την τροπολογία 11, α, καταπίπτει. Άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 4, 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το 2 έχουν τροπολογία 12. Ελίζαμπε Σρέντες, γιατί είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 έχει αποσυρθεί και ψηφίζουμε πλέον το σύνολο της ούτως τροποποιητή εκθέσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 30 ψήφι πέρα. 4 κατά 0 αποχές. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά πάντα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 1, 0 συγγνώμη αποχές. Και σας ευχαριστώ. Οπότε περνάμε στο σημείο 20. Πρόκειται για το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή ΙΜΚΟ επί της έκθεσης για μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης της Γιούτα Steinrock. Παραγραφός 1. Συμβιβαστική α τριών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας και λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συμβιβαστική β τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβαστική C 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 4 ε, τροπολογία διαγραφής 10 της Αρίας Αία υπέρ κατάργησης της παραγράφου 4 κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 4 συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 5, συμβαστική ε, ε, υπερκατάποχες εγκρίνεται. 6, ε, συμβαστική F, ε, υπερκατάποχες εγκρίνεται. Παραγραφός 5, τροπολογία 18 της συγκήτριας και της Μπερναδετ Με έτοιμα ψηφοφορίες κατά τμήματα. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα λοιπόν, κατά οι αποχές απορρίπτεται νομίζω να το επαληθεύσουμε όμως άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 18 Tout le monde a Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα, αλλά περιλαμβάνει μια προφορική τροπολογία. Έχει κάποιο αντίρρηση για την προφορική όχι. Δεύτερο τμήμα λοιπόν όπως τροποποιείται, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τροπολογία 23 Μαρτιν Κάσλερ υπέρ κατά αποχές εγκρινέται τροπολογία 24 της Γιώτα Στάινρου και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρινέται τροπολογία 25 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία Ψήφισαν άπαντε πέρα τη ψηφοφορία. 31 υπέρ, 4 κατά, 0 αποχέ. Συγχαίρουμε την εισηγητρία. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία που είναι η ψηφοφορία για τις τροπολογίες που θέλουμε να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ε, για την εξέταση ταυτόχρονα του Γενικού Προγράμματος ε, REFIT συμπεριλαμβάνοντας ε, την ανακοινωσή της 2-3 Οκτωβρίου της Κομισιόν για το ίδιο θέμα μετά την παραγραφό 5 τροπολογία 1 των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 1 ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας 27 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται δεν χρειαζόταν επαλήθευση. Παράγραφος 5. Ε, τροπολογία 2. Με προφορική τροπολογία. Αντίρρηση για την προφορική. Όχι υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 10, τροπολογία 4, ίδιας σοσιαλιστών υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, μετά την παραγραφό 10, τροπολογία 5, τον νησιά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 11, τροπολογία 6, των σοσιαλιστών υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 11, τροπολογία 7 των πρασίνων, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 7 των πρασίνων. Ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 18 κατά. Πράγματι απορρίπτεται. Παραγραφός, μετά την παραγραφό 12, τροπολογία 8 των σοσιαλιστών υπερκατά αποχές εγκρίνεται ίδια παράγραφος, ε, παράγραφος 1, 9 ε, των σοσιαλιστών υπερκατά αποχές απορρίπτεται. Στο τμήμα 2 της ίδιας παραγράφου 10 των σοσιαλιστών κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι 4 της ίδιας παραγράφου, 11 τροπολογία των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρινέται. Παράγραφος 12 μετά το εδάφιο 4 τροπολογία 12 το ECR με έτοιμα ε, να ψηφίσουμε κατά τμήματα πρώτο τμήμα μέχρι το particularly ποιος είναι υπέρ για αυτό το πρώτο τμήμα κατά αποχές Ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Το πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Για το πρώτο τμήμα εγκρίνεται με 20, 15, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην παραγραφό 12, 5, 13 των σωσιαστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 12, τροπολογία 14 του ΙΣΕΑΡ υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε άρχεται η επαλήθευση για την τροπολογία 14 ψήφισαν άπαντες της ψηφοφορίας 7 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται σαφώς τροπολογία 15 σοσιαλιστών με προφορική τροπολογία Συγγνώμη. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 15 χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της ίδιας ομάδας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 της ίδιας ομάδας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 της, του ECR μετά την παράγραφο 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ολοκληρώσαμε αυτές τις τροπολογίες που θα υποβληθούν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες και θα πάμε προς τα πίσω διότι θα πάμε τώρα στο σημείο 11 όπου θα εξετάσουμε την έκθεση πρωτοβουλία του πώ μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντο για τη δημιουργία θέσεων εργασία σε επιχειρήσει και νεοσύστατε επιχειρήσει. Πρόκειται και το σχέδιο έκθεση τη συναδέλφου μα, Ανθέα Μακεντάιερ, όπου θα εξετάσουμε τις 276 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας, όπως ξέρετε, για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός φιλόξενου πλαίσιου εργασίας για τις επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που ξεκινάνε για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες σας. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Υπήρξαν 276 τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες. μόνο μία παράγραφος από όλη την έκθεση δεν έχει ε, προταθεί να τροποποιηθεί. Και αυτό μάλλον ε, ε, οφείλεται στο ότι μόνο εγώ ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα CREATE, που νομίζω ότι είναι σημαντικό παρόλα αυτά. Μερικές παράγραφοι υπέστησαν έως και εννέα τροπολογίες. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο συμβιβασμών, γιατί φυσικά δεν θέλουμε να ψηφίσουμε 276 τροπολογίες. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα υπάρξει συμφωνία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υποβλήθηκαν τόσες τροπολογίες και Χαίρομαι επίσης ε, για το πνεύμα συνεργασίας ε, που διαπιστώνω μέσω των τροπολογιών. Υπάρχουν ε, πολλές από αυτές που με χαρά θα υποστήριζα. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα. Ε, το τεστ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι πρώτα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα δημιουργήσουμε μικρές επιχειρήσεις, πώς τους επαχθέστερους, τις 10 επαχθέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις θα τις ελαφρύνουμε. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ήδη λάβαμε δύο γνωμοδοτήσεις για το θέμα αυτό και όλα αυτά βοηθάνε. Άρα η πρόκληση ενώπιόν μου είναι να δημιουργήσω, να καταλήξω σε συμβιβασμούς με τους οποίους να μπορούν να συμβαδίσουν όλοι και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Θα πρέπει να κάνουν συμβασμούς για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση πώς θα συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση επιχειρηματικότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα, χρηματοδότηση από την Ένωση, γυναίκες ε, επιχειρηματίες και υγεία και ασφάλεια. Για τους υπόλοιπους συμβασμούς θα βασιστούμε στο υπάρχον κείμενο. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει αντί να είναι μακροσκελέστατος ένα συμβασμός θα μπορούσαμε να ε, κατατμήσουμε τις παραγράφους θα συνεργαστώ με όλους τους κοιόδης, θα κυκλοφορήσουν οι προτάσεις μου πριν από την επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών που ελπίζω ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα είτε τη μεθεπόμενη. Προσβλέπω λοιπόν στα σχόλια όλων ημών ε, για τις τροπολογίες που έχουν ήδη υποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Μπένιον. Α, όχι, καλύτερα πρώτα ο κύριος Θέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη συζήτηση την ξεκινήσαμε χθε με το REFIT, REFIT. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει εξέτασης γιατί η δημιουργία ενός φιλόξενου για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος είναι η πιο ασφαλής οδός για δημιουργία θέσεων εργασίας, κάτι που είναι άκρος απαραίτητο στην Ευρώπη. Όμως και εδώ, όπως και οπουδήποτε αλλού στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε ανοιχτά και τα δύο μας μάτια και να περπατάμε και με τα δύο πόδια. Ούτε μονόφθαλμοι να είμαστε, ούτε κουτσί. Και γι' αυτό θα πρέπει να ε, συνδυάσουμε την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζονται επιχείρηση, αλλά και την ε, ασφάλεια ε, που επιβάλλει και η νομολογία του δικαστηρίου. Θα έλεγα λοιπόν στην κυρία Μάκιντάρ ότι διάβασα πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες της δικής μου πολιτικής ομάδας που έχουν ως στόχο να μην υπάρξει ε, ανατροπή τη ισορροπίας προ τη μία ή την άλλη όψη νομίσματο. Θα ήθελα να πω ότι έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, κάποιες αφορούν ε, ε, διατάξεις οδηγίας για την εργασία και ήταν επικοδομητική η διάθεσή μου. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μάκητα να προσπαθήσει να καταλάβει ότι ήδη στην ιστορία του Κοινοβουλίου έχουν ε, γίνει πολλές προσπάθειες. Έχουμε σημαντικούς συμβιβασμούς και 15 Μαΐου του 12 είχαμε ε, συμπεριλάβει πάρα πολύ σημαντικές διατάξεις με μείωση του άκθους για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί περιλαμβανόταν ένα δόγμα πολύ σημαντικό και υπήρξε συμφωνία. Ποια ήταν η συμφωνία? Ότι το διοικητικό άχθος δεν θα πρέπει ε, να το καταργήσουμε σε σημείο που τελικά τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, και της αξιοπρεπούς εργασίας ε, να καταρριφθούν. Ε, φαντάζομαι θα το καταλάβει η κυρία Μακιντάιρ. Θα κάνουμε τη μέγιστη αντιπροσπάθεια, χωρί όμω να θέσουμε σε κίνδυνο τα πρότυπα και τους κανόνες του κανόνε του Διεθνού Γραφείου Εργασία και τη αξιοπρεπού εργασία εν γέννη. Διότι, κυρία Μακιντάιρ, υπάρχει αντίφαση μεταξύ ε, των επιχειρήσεων, των χρημάτων, τη υγεία των εργαζομένων Εμείς ε, θα έλεγα να σας πω ότι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, κυρία Μακιντάρε, το κέρδος και την επιχείρηση, την επιχειρηματική δραστηριότητα, αν αυτό έρχεται σε βάρος της υγείας των εργαζομένων. Η κυρία Γκουτιέρεθ Πριέτο και εγώ υπογράφουμε μια τροπολογία πάρα πολύ σημαντική που είναι και κόκκινη γραμμή της ομάδας μας αν θέλετε. Δηλαδή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αποσυνδέοντας ε, ή μάλλον ε, καταργέντοντας αυτή την αναφορά. Και αν μιλάμε για ωράριο εργασίας, working time, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ελαστικό. Πρέπει να πούμε ότι εξακολουθούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια οδηγία, από το 2003 την περιμένουμε, που θα έπρεπε ουσιαστικά και να επιλύσει τα ζητήματα τα οποία έχει επισημάνει το δικαστήριο και λέει ότι πρέπει να ε, λυθούν στο σώμα του κειμένου αυτού που έχουμε. Υπάρχει ασυμμετρία μεταξύ αυτών που λέει η οδηγία και αυτών που αποφάσισε στην δημιουργία του δικαστήριου και που πρέπει να τη σεβαστούμε. Θα ήταν ε, λοιπόν ε, ρηψοκίνδυνο να διαγραφεί, να γίνει απόπειρα να διαγραφεί ε, διατάξει όπως είναι αυτή για την προσωρινή εργασία. Δεν μπορούμε έτσι με μία μονοκοντιλιά να σβήσουμε μία ολόκληρη οδηγία. Πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μία αρμονική σύνθεση. Κύριε Μακιντάρη, σας εγγυώμαι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αναζήτηση συμβιβασμών, αλλά σας λέγω ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για τη δική μας ομάδα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων και δει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω τον λόγο στον Φιλμπάνιαν να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών ότι οι ψηφοφορίες μας ήταν πιο σύντομες, ε, έγιναν πιο, δυσκο... πιο γρήγορες από ό,τι είχαμε προβλέψει. Βλέπω λοιπόν ότι πολλοί βουλευτές ε, που ενδιαφέρονται για τους φακελούς που θα εξετάζουμε στη συνέχεια δεν βρίσκονται εδώ. Για να μην αλλάξουμε λοιπόν τη σειρά των εργασιών μας, σας παρακαλώ να ενημερώσετε τα μέλη σας ώστε να έρθουν εδώ. Δίνω το λόγο στον Φιλμπένιαν. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εκ μέλους του Φίλιπ Ντεμπάκερ που δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Ο Φίλιπ θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για τη δουλειά της σε αυτό το φάκελο, για τις δηλώσεις ότι πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Ε, ο Φίλιπ πιστεύει ότι μιλήσαμε αρκετά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβουμε ε, δράση για να υποστηρίξουμε τους επιχειρηματίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χαράξει πολιτικές ώστε να βοηθήσει κατά προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει υποβάλει ο Φιλίπ κάποιες τροπολογίες για τη βελτίωση της χρηματοδότησης με εφόρο τρόπο όχι με βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά με νέε μεταρρυθμίσει για την προσέλξη νέων επενδυτών και κεφαλαίων, με εκπαιδευτικά συστήματα, με καταρτισμένους εκπαιδευτικού προσαρμοσμένου στι επιχειρηματικέ ανάγκε με ταυτόχρονη συμπεριλήψη της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα τρίτων, μείωση του διοικητικού άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και για τις μεγαλύτερες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν αποτελεί προς το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης μια ευέλικτη αγορά με ένα δίκτυο ασφαλείας, η ισορροπία ε, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερο εργατικό δυναμικό στην αγορά. Ο Φιλίπ ε, προσδοκεί να συζητήσει τις ε, τροπολογίε μας τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Σέζιο Κουτέρες. Και υπάρχουν και άλλοι που θα ήθελαν να παρεύουν για την εκθέση της κυρίας Μακεντάρ. Όχι. Σέζιο Κουτέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες, τις 276 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το σχέδιο έκθεσης και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ κοινοί παρονομαστές. Αν γίνει λοιπόν προσπάθεια από την εισηγητερία, πιστεύω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, κυρίως για να εστιάσουμε στα προβλήματα που πραγματικά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή χρηματοδότηση, πρόσβαση στην πίστοση, σε πιστώσεις πρέπει να είναι βιώσιμη για όλες τις επιχειρήσεις και βραχυπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα η χρηματοδότηση αυτή. Επίσης, απλούστευση των ευρωπαϊκών κανόνων και των κοινοτικών κανόνων για να ε, ενισχυθεί η ενιαία αγορά. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία εάν η συγγήτρια ε, εγκαταλείψει κάποια θέματα που και προβλήματα δημιουργούν αλλά και δεν έχουν καμία σχέση κατά την άποψή μου με τα προβλήματα των ε, επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασία και για άλλα ζητήματα. Όπως ε, σχολίασε ο συντονιστής ε, της Σοσιαλιστική ομάδας, ό,τι έχει να κάνει με την οδηγία σχετικά με το ωράριο εργασίας και άλλες οδηγίες που πιστεύουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την γραφειοκρατία, με την απλούστευση, αλλά με απώλεια δικαιωμάτων ε, τελικά. Και αυτό είναι άλλη συζήτηση, άλλο θέμα. Δεν είναι για αυτή την έκθεση. Η σοσιαλιστική ομάδα έχει καταθέσει τροπολογίες διαγραφής ε, από κοινού με τους Πρασίνους ε, και κάποιον άλλο βουλευτή Ακριβώς για αυτές τις τροπολογίες θέλω να σας πω, επειδή θεωρούμε ότι άλλο η απλούστευση γραφειοκρατίας και άλλο απόλυτα δικαιωμάτων, μεγάλο χάσμα υπάρχει, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτή τη στιγμή και επίσης οποιαδήποτε βελτίωση θα μπορούσε ε, να είναι υπέρ των μικρών ε, και των μεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να εγγυάται και τα ε, εργασιακά δικαιώματα. Συμφωνούμε με πολλέ ε, τροπολογίε, επιχειρηματική κουλτούρα, βελτίωση απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση κτλ. Υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας πολύ σημαντικά, απλά ε, θα χρειαστεί η συγκέντρια όταν προτείνει συμβιβασμούς, επειδή βέβαια υπάρχουν πάρα πολλέ τροπολογίε. αν λοιπόν η συγκέντρια κάνει μια παραπάνω προσπάθεια για να αποσύρει ορισμένα ζητήματα που είναι επίμαχα για την Επιτροπή Απασχόλησης. Προσωπικά θα σας προσφέρω τη συνεργασία, την οχήρα συνεργασίας προς εσάς για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και για να συντάξουμε μια καλή έκθεση που έχει καλά στοιχεία, έχει εύστοχα σημεία αλλά και λάθη, έχει σφάλματα γιατί περιλαμβάνει θέματα που κατ' δεν πρέπει να είναι στο θεματολόγιο της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρέμβει η Κομισιό. Κύριος Πεντούτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Έχουμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Παραμένουν όμως ε, δύο σημεία που μας ανησυχούν. Πρώτον, το ζήτημα των επενδύσεων που δεν έχουν αποδόσεις και το ζήτημα της απασχόλησης. Διότι επικίνδυνο να έχουμε ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς ε, μείωση της ενεργείας. Γι' αυτό το λόγο το ζήτημα των επιτροπών πλαισίων που θα επιτρέπουν στις ε, μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ευρώπη είναι, ε, έχει όλο και πιο κρίσιμη σημασία. Να επισημάνω ότι εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του επόμενου Φεβρουαρίου που θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική πολιτική, η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα θέμα που αφορά και αυτό το πλαίσιο για τις επενδύσεις και για την μείωση της ενεργείας. Κύριε Συγγήτρια. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την πολύ θετική του συμβολή. Θα ήθελα να καθησυχάσω τις ανησυχίες ότι προσπαθώ να καταργήσω την νομοθεσία περιγείας και ασφάλειας. Στην παράγραφο 25 μάλιστα, για την οποία προτάθηκαν αρκετές τροπολογίες, ορίζω την στρατηγική υγείας και ασφάλειας. Ο στόχος μου είναι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Για ποιο λόγο για να επιτύχουμε καλύτερο επίπεδο πρόληψης και καλύτερο επίπεδο συμμόρφωσης. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο να ε, καταλήξουμε σε συμβιβασμό σε αυτό το τομέα. Δεν θα σας εκπλήξει ότι θέλω να διατηρήσω την παραγραφό μου αυτή. Ε, ε, δεν μπορώ να υποστηρίξω λοιπόν τις ε, τροπολογίες για διαγραφή, αλλά δεν είναι πολλές. Στο σύνολο τους οι τροπολογίες είναι πολύ θετικές και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα εξετάσουμε τις εμβιβαστικές τροπολογίες της 17 για να τις ψηφίσουμε στη συνέχεια. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σημείο της μεσής δίδαξης και περνάμε στο σημείο 22. όπου θα εξετάσουμε το σχέδιο απόφασης για την ενισχυμένη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Θα εξετάσουμε τις 50 τροπολογίες που υποβλήθηκαν για το σχέδιο εκθέσης του Φρεντρικ Νταρντέν και του δίνω το λόγο. Merci, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι θετικός εναντί αυτής της πρωτοβουλίας της Επιτροπής που θέλει να κάνει επίσημη την ανεπίσημη προσπάθεια που κάνει για την ε, συγκριτική ε, κατάρτιση. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, ορισμένες τις έχω κάνει και εγώ. Και για να συμπληρώσω λοιπόν έκανα αυτές τις τροπολογίες στην αρχική μου ε, σκέψη. Και για τις ε, άλλες τροπολογίες έχω γενικά θετική άποψη. Θα τις συγκεντρώσω γύρω από κάποια ενοιολογικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι μέλη αυτού του δικτύου. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, η νομοθετική αρμοδιότητα είναι σε υποεθνικό επίπεδο. Άρα Πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη εκπροσώπηση αυτού του επίπεδου αρμοδιότητε, αλλά το δίκτυο να μείνει όχι πολύ εκτεταμένο, αποτελεσματικό και κάθε κράτο να έχει ε, μία ψήφο με πλήρη δικαιώματα για λόγους ισοτιμίας. Ήδη το συζήτησα με τον κύριο Μπέκερ θα μπορούσαμε ίσως ε, να βασιστούμε και να εμπνευστούμε σε αυτά που έγιναν για την πρωτοβουλία για τους νέους όπου υπήρξαν δυσχέρειες αλλά τις ξεπεράσαμε. Δεύτερο θέμα, ποιοι άλλοι θα συμμετάσχουν εκτός από τις ε, δημόσιες ε, τους δημόσιους οργανισμούς ε, απασχόλησης πρέπει να είναι επιθεώρηση εργασίας, άλλοι κοινωνικοί εταίροι, πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν και αυτοί για να αποφεληθούμε από την πείρα τους, χωρίς όμως να επιβαρύνουμε τη λειτουργία, ίσως θα μπορούσαν να είναι παρατήρητες. Και επίσης πρέπει να συνεργαστεί με κάποιους άλλους φορείς το δίκτυο αυτό. Η Κομισιόν δεν είπε τίποτα από αυτόν, εμείς ε, καταλήξαμε σε κάποιο κατάλογο όπου αναφέρονται και ιδιωτικοί φορείς, βεβαίως βάση θα είναι οι δημόσιοι οργανισμοί απασχόλησης. Αλλά βεβαίως πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί οι ιδιωτικοί φορείς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Πέρα λοιπόν από τα μέλη και τους συνεργαζόμενους φορείς, πώς θα υπάρξει η θεσμική κατανομή αρμοδιοτήτων και η κατεξοδότηση πράξη. Και εδώ υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις που φαίνονται από τις τροπολογίες, γιατί ορισμένες τροπολογίες θέλουν να καταργήσουν τη διαδικασία έγκρισης της μεθοδολογίας και των δικτών μέσω κατεξοδότηση πράξεων, να δούμε εδώ τι θέση ε, θα έχει η Επιτροπή μας. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει άποψη του Κοινοβουλίου. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εκτελεστικές πράξεις υπερβολικές. Αν καταργήσουμε την κατεξοδότηση νόμος ε, πράξη, θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική μέθοδος για να προτείνουμε δείκτες. Ποιος θα το κάνει εμείς. Πρέπει να λάβουμε θέση. Αλλά πέρα από τη δική μας θέση θα το συζητήσουμε σίγουρα και στον τριμερή διάλογο γιατί το Συμβούλιο μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Να λοιπόν μερικά κέντρα βάρους που θα προκαλέσουν συζήτηση. Ήδη το εξετάζω το θέμα για να εκπονήσω συμβιβασμούς που θα είναι διαθέσιμοι για την ψηφοφορία στις 5 Δεκεμβρίου για να ψηφίσουμε στις 9. Και είμαι στη διάθεση των σκιωδών για να συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές. Μεθαύριο θα συναντηθούμε για το στόχο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπέκα. Μετά ο κύριος Ευχαριστώ. Εισαγωγικά να πω ότι έχω πολύ θετική στάση για την εργασία του εισηγητή με πολύ ευσυνείδητο τρόπο. Αντιμετώπισε περίπλοκα θέματα, όπως μας τα παρουσίασε, τη σχέση των δομών με τα κράτη-μέλη, με τους ενιαίους ευρωπαϊκούς στόχους. Πολύ θετικά αντιμετωπίζω γιατί κάποιες όχι πολύ, κάποιες όχι πολύ σαφώς ε, διατυπωμένες σκέψεις της Επιτροπής μας επέτρεψαν παρόλα αυτά να καταλήξουμε σε θετική στάση και μπορώ να σας πω ότι μπορώ να εκφράσω τη θετική γνώμη του ΕΛΚ. Τονίζω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο των δημοσίων οργανισμών απασχόλησης όπου όμως θέλουμε να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς. Υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες εξέβρεση εργασίας. Υπάρχουν περιφερειακές δομές, δεν είναι πάντα εθνικές. Και όπως μας είπαν οι οργανισμοί απασχόλησης εδώ και χρόνια, υπάρχει ήδη ένα δίκτυο των οργανισμών απασχόλησης που λειτουργεί άτυπα αλλά επιτυχώς. Γι' αυτό ήθελα οπωσδήποτε να μην ε, θέσουμε εμπόδια σε αυτή τη λειτουργία που ήδη υπάρχει. Και στη συζητήσεις με τον εισηγητή και άλλους ε, είδα ότι έχουν θετική στάση. Θεωρώ ότι θα είναι δυνατόν ε, οι διάφορες δομές που έχουμε για να αυξηθεί η απασχόληση στην Ευρώπη να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. Γιατί τα διάφορα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη καταφέρει να έχουν τις κατάλληλες δομές. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία της Κομισιόν και ευχαριστώ πολύ. Ο Φιλ Μπένιον και μετά ο Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω είναι χρήσιμη συμβολή της Κομισιόν. Θα συμπεριλάβει νέες δομές θα ενισχύσει τις φυστάμενε. άρα καλοδεχούμενη πρόταση της Κομισιόν. Ε, έχω κάποιες ελάχιστες τροπολογίες, ε, ε, κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι θα πρέπει να μειωθεί η ανεργία των νέων. Το δίκτυο θα πρέπει να θεσπίζει και να οδηγήσει, σε ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών για την κατάρτιση, επαγγελματική εκπαίδευση, όλε αυτέ τι ανάγκε και τα μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέου να αποκτήσουν τι απαραίτητε δεξιότητε για να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασία. Επίση η μαθητεία ε, και η απασχόληση συνδυαζόμενη με κατάρτιση είναι σημαντικέ πτυχέ. Το δίκτυο θα πρέπει επίση ε, με τι ιδιωτικέ υπηρεσίες απασχόληση να συνεργάζεται για να αναγνωριστούν διαφορέ μεταξύ των συστημάτων και μοντέλων απασχόληση των κρατών μελών και για να είναι πιο αποτελεσματικέ οι προτάσει σε κάποια κράτη-μέλη. Και έρχομαι σε αυτά που ο κύριο Μπέκερ. Επίση, το σύστημα θα πρέπει να εντοπίζει ε, χάσματα και κενά στι δεξιότητε, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ε, μέτρα τα κράτη-μέλη για να γεμίσουν τα κενά αυτά. Και σε ό,τι αφορά τα αρχικά σχόλια τη ηγητή, συμφωνώ και προσβλέπω στη συνεργασία μα για τη ε, διατύπωση συμβαστικών τροπολογιών. Jean Lambert, puis Thomas. Jean Lambert και μετά Thomas Mann. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Νταγντά ε, για τη δουλειά του και περιμένω και εγώ με ανυπομονησία να συζητήσουμε κάποιες συμβαστικές τροπάσεις. Ε, καταθέσαμε λίγες τροπολογίες, διότι κατά εμάς υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν κάποιες οργανώσεις σε κάποια δίκτυα, ε, παραδείγματος χάρη σχέση, διασύνδεση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ανέργους. Και νομίζω ότι κάποιες προτάσεις για το τι γίνεται, τι συνεργασία υπάρχει με τις τοπικές περιφερειακές αρχές. Χρήζει κάποια συζήτηση, σηκώνει συζήτηση διότι ναι μεν είναι σωστή ανάλυση ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση στο σύστημα και θα πρέπει αυτό να λαμβάνει υπόψη και στο δίκτυο. Απ' την άλλη, είναι σημαντικό όταν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά να δούμε από ποιες άλλες ε, γύρω-γύρω έτσι ο οργανός μπορεί να αντλήσει το δίκτυο για να μην υπάρξει αλληλεπικάλυψη εργασιών. Αφού έχουμε να κάνουμε και με ένα νομικό κείμενο. Η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι όχι να φορτώσουμε αυτό το νομικό κείμενο με στοιχεία που θα πρέπει μετά να αποτελούν κανόνε για τα επόμενα 6-7 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ανεργία και την απασχόληση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί το θέμα να μην είναι ε, μείζον. Υπάρχουν άλλοι τομεί ε, του πληθυσμού ή ομάδε ε, που. Ε, που εκπροσωπούνται. Δεν είναι μόνο οι νέοι δηλαδή στου οποίου εστιάζουμε, αλλά μπορεί να είναι άλλε κατηγορίε πληθυσμού που είναι εκτό τη αγορα εργασία, σε κάποια κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να διατυπώσουμε προτάσεις ε, για να καλύψουμε, ε, να λάβουμε υπόψη μα αυτέ τι διαφορέ. Πάντως θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή για την εξέβρεση συμβασμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις θετικές εκτιμήσεις ε, των προηγουμένων. Πολύ καλή δουλειά, Φρεντρίκ. Θαυμάσια. Και επειδή τέθηκε το ερώτημα εάν το ΕΛΚ θα στηρίξει, νομίζω ότι μπορεί να στηρίξει με βάση την πύρα που έχουμε και στην Αυστρία. Έχουμε καλή πύρα, καλή εμπειρία με, τις, ε, με τους δημόσιους οργανισμούς ε, απασχόλησης. Αλλά υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι καθόλου δεν είναι στην κρίζα εργασία, είναι κανονικές επιχειρήσεις, κανονικές ε, ε, λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά βέβαια πρέπει να ελέγχονται. Η συνεργασία είναι το σημαντικό. Και δεύτερο, έχει απόλυτο δίκιο η Jean Lambert πρέπει να ασχοληθούμε βεβαίως με τους νέους, είναι η προτεραιότητά μας, η πρωτοβουλία, τα έξι η εγγύηση, είναι πολύ σημαντικά μηνύματα που θέλουμε να αποστείλουμε, αλλά για τις δημόσιους οργανισμούς απασχόλησης υπάρχουν και άλλες ομάδες με τις οποίες πρέπει να απασχοληθούμε, να τις ε, καθορίσουμε συγκεκριμένα, να τις οριοθετήσουμε, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη αρκετά αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, στην 62 τροπολογία λες ότι δεν θέλεις να υπάρχει ιεράρχηση. Αλλά το θέμα δεν είναι πρώτα να έχουμε στόχους, αλλά να βοηθήσουμε και μέσω μιας κοινή μεθοδολογίας. Γιατί δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται θέμα ε, ιεράρχησης. Βεβαίως να πούμε πρώτα οι νέοι, μετά οι γυναίκες, μετά οι μακροχρόνια άνεργοι. Γιατί λοιπόν έχει υποβάλει αυτή την τροπολογία. Κατά τα υπόλοιπα δεν έχω πρόβλημα και σίγουρα μεταξύ των σκιωδών θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον Φρέντρικ. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλος συναδέλφο που θα θέλει να παρέμβει. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί το λόγο. Η Κομισιόν θα ήθελε να πει κάτι. Δεν έχει να πει κάτι η Κομισιόν. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σιγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους διάφορους προλαλήσαντες ε, για τα ευνοϊκά του σχόλια για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και είμαι ακόμα πιο πεπισμένος μετά από αυτές τις ε, παρεμβάσεις ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς που θα βοηθήσουν στην πρόθεση του σχέδιου της Κομισιόν και αυτού του σχεδίου έκθεσης θα ήθελα να επανέλθω για μια στιγμή σε αυτά τα θέματα, στις αποστολές, ε, θα έλεγα, αυτού του δικτύου. Είναι σαφές ότι η καταπολέμηση της ενεργείας των νέων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους άλλους ε, στόχους, τα άλλα, τις άλλες ομάδες, τις άλλες κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν επίσης από την ανεργία. Και σήμερα ισχύει... αυτό που ισχύει είναι ότι σε ορισμένε χώρε ισχύουν κάποια πράγματα που δεν ισχύουν σε κάποιε άλλε και ότι τα πράγματα αυτά δεν θα ισχύουν για πάντα. Πρέπει να επιμένουμε λοιπόν σε μια αναγνωρισμένη προτεραιότητα σήμερα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων αλλά να μην στοχεύουμε μόνο αυτού του είδου την ανεργία. Θα πρέπει να ανοιχτούμε και στι άλλε ομάδε του πληθυσμού, φυσικά με μια λογική ορισμού προτεραιοτήτων ε, που πιστεύω θα πρέπει να ενσωματωθεί στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έτσι θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες τους συμβιβασμούς. Δεν θέλετε να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα του Τόμας Μάνου. C'était le 62. 62, λέει ο κ. Στουμάνου. Oui, par rapport à cet Ναι, σε σχέση με αυτή την τροπολογία, την 62, που αντιστοιχεί σε κεψέντρες που άκουσα από την Επιτροπή των Περιφερειών στο πλήσιο των συζητήσεων ε, που είχαμε επί του θέματος ε, με είχαν καλέσει μια συζήτηση πιστεύω ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε μια λογική ανταγωνισμού μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και μια λογική ε, αξιολόγηση των επιδόσεων των μεν σε σχέση με τον δε. Γι' αυτό έχουμε αυτή την τροπολογία. D'accord. Euh, donc, nous en Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα προτείνει κυρίως ο κύριος Ηγετής στις 5 Δεκεμβρίου ώστε να ψηφίσουμε στην έκτακτη συνεδρίασή μας στις 9 Δεκεμβρίου. Ολοκλώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο σημείο 23 όπου θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που συντάσσουμε για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σε σχέση με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012. Δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Άνταμ Κώσα, για την εξέταση των 31 τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Κύριε Σίγητα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αληθεύει, όπως είπατε, 31 τροπολογίες βλήθηκαν για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Τρία μέλη υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήρια εκ μέρους των Πρασίνων η κυρία Λάμπερτ και εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Σίπερ. Και εγώ επίσης υπέβαλα δύο τροπολογίες. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά καλά σε σχέση με το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Ε, προχωράμε αρκετά γρήγορα, διότι έγινε η συνάντησή των σχεδόν που εξετάσαμε όλες τις τροπολογίες και ουσιαστικά δεν υπάρχουν προβλήματα. Όλες οι τροπολογίες, πέραν μία ή δύο, δεν παρουσιάζουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντιθέτω, έχουμε καταλήξει σε δύο συμβαστικέ προτάσεις ε, βάσει των οποίων όπως φαίνεται θα έχουμε τη συμφωνία των ομάδων την επόμενη φορά που θα το εξετάσω όλο αυτό σε πιο βάθο. Υπάρχουν ε, ε, δύο τροπολογίε που θα ήθελα να εξετάσω σε περισσότερο βάθος τώρα. Η ομάδα των Πρασίνων μου ζήτησε μια προφορική τροπολογία. Αναφέρομαι στην ε, τροπολογία αριθμό 15 και από ό,τι άκουσα θα γίνει δεκτή διότι ουσιαστικά αναφέρεται στην ίση μεταχείριση και τονίζει τη σπουδαιότητά της ε, και με για μια ισότιμη μεταχείριση. Και μετά υπάρχει μια άλλη τροπολογία που προσφέρει κάποιο πρόβλημα για μένα. Ίσως θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Πρόκειται για τροπολογία 22 της ομάδας των σοσιαλιστών. Κατανοώ την πρόθεση στην οποία στηρίζεται η τροπολογία αυτή και πιστεύω ότι απουσία ουσιαστικά αρμοδιοτήτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια από τα βήματα εδώ πέρα και αυτό με ανησυχεί. Επίσης υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο πιστεύω θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αναφέρομαι στην τροπολογία 30 όπου μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, γίνεται αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Χρειάστηκε να κοιτάξω σήμερα το πρωί τη συνθήκη. και θα το χαρτί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γίνεται αναφορά στον κοινωνικό χάρτη εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσω να υποστηρίξω την τροπολογία 30. Από τις 31 λοιπόν τροπολογίες είναι βέβαιο ότι ήδη μπορώ να υποστηρίξω τις 29. Και όπως ανέφερα προηγουμένως έχουμε συμφωνήσει και για δύο συμβέσμους Έχει διευκρινιστεί λοιπόν ε, η πρόθεση που, στην οποία στηρίζεται η καθροπολογία και έχω μια σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή ότι όντως προσθέτουν αξία. Και είμαι βεβαίω ότι και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορέσει να τις ε, λάβει υπόψη κοιτάμε, ζητήματα κοινωνικά και απασχόλησης. Ε, και αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Birgit Sibel και Jean Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ θερμά τον κύριο Κόζα για την ε, ετοιμότητά του να συνεργαστεί σε αυτό το θέμα και επιβεβαιώνω ότι οι τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν ε, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο δυσχεριών στην περαιτέρω συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη βασίζονται στην αρχή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πολύ βασική αρχή, είναι αδιέρετα και για τον τομέα της απασχόλησης, γι' αυτό ασχοληθήκαμε με κάποια συγκεκριμένα θέματα. Να αναφέρω μόνο ορισμένα από αυτά που προκύπτουν από τις τροπολογίες μας. Πρώτα απ' όλα βέβαια είναι το θέμα του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε, η αυτονομία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όλα αυτά πρέπει να μην φυγούν. Επίσης το θέμα της ε, ελεύθερης διακίνησης ε, των εργαζομένων στην Ευρώπη είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης και πρέπει επειδή περνάμε δυσχερείς περιόδους ε, να διατηρηθεί αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να το πούμε σαφώς αυτό Επίσης να αναφερθούμε και στις διακρίσεις, να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις. Ε, ποτέ δεν σταματάει αυτό το καθήκον. Θα ήταν σκόπιμο επιτέλους το Συμβούλιο να εγκρίνει την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Επίσης, ευχαριστώ τον εισηγητή, γιατί από ό,τι φαίνεται θα υποστηρίξει την τροπολογία μας 30 για την 22 Σίγουρα στην επόμενη συζήτηση θα τα ξαναπούμε. Και μία ερώτηση στον εισηγητή για την τροπολογία μας 14. Χθες ε, του προτείναμε μία νέα διατύπωση. Σας τη στείλαμε. Αν μπορείτε να τις ρίξετε μια ματιά, σας παρακαλούμε συντόμως να μας πείτε αν ε, αυτή η αναδιατύπωση μπορεί να γίνει δεκτή από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την ε, προθυμία του να λάβει υπόψη του τις ε, κατατεθήσεις τροπολογίες. Επιβεβαιώνω ότι σε ό,τι αφορά την τροπολογία μας παρθμών 15 θα δεχθούμε αυτή την επιπλέον αναφορά Επίσης θα συζητήσουμε, όχι ουσιώδης βέβαια, ως ε, ε, σημασίας τροποποίησης για τις τροπολίες 18, 19 και άλλη μία νομίζω, όπου ε, είχαμε ξεκινήσει με ένα κομμάτι του κειμένου μια έκθεση επιτροπή μα, αλλά θα θέλατε να το χρωματίσετε διαφορετικά. Θα το συζητήσουμε ευχαρίστω μαζί σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Επιτροπή απασχόληση ε, συμβάλλει ε, φέτος ε, στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την τροπολογία 22. Συντονισμός κοινωνικής ασφάλισης. Έχω εμπειρία γιατί έχω εργαστεί για κάποια χρόνια στο θέμα αυτό. Επειδή έχουμε συζητήσει και τα επιδόματα ενεργείας, φαντάζομαι ότι σε αρκετά κράτη-μέλη υπάρχει εντύπωση θα πρέπει να υπάρξει παράταση από τους τρεις στους έξι μήνες. Αυτό έτσι λίγο ε, ε, είναι μετέωρο στα κράτη-μέλη, συζητείται ενδεχομένως ε, αυτό το καιρό. Θα ήταν καλό να δώσουμε και εμείς ως Επιτροπή ένα ισχυρό μήνυμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόεδρος, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν τον λόγο. Όχι. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουδής. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Όχι, μάλιστα. Άρα, κύριε Σιγητά, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε, αν θέλετε, στις παρεμβάσεις και ιδίως στην κυρία ε, Ζίπελ για την τροπολογία 14. Έχετε το λόγο. Κύριε Σκόζα, σας ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές. και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι όλες οι παρεμβάσεις ε, κινούνται ε, στο ίδιο μήκο Βέβαια κάποιες έθεσαν πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ετέφει το ζήτημα των οριζόντιων οδηγιών από τους σοσιαλιστές. Ως άτομο με αναπηρία φυσικά και δεν μπορώ παρά να στηρίξω απόλυτα την ιδέα για μια οριζόντια οδηγία. Βέβαια θα ήθελα να αναφέρω το εξή. Θα πρέπει να προχωρούμε σε συνάρτηση με τις αρμοδιότητες που ανατίθεται σε επιτροπές. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη βασική ιδέα. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 14, ε, σας ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα να αναφέρω στην ε, πρώτη μου παρέμβαση ότι μπορώ να δεχθώ τις προτάσεις για την τροπολογία 14 Άρα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν αυτό το ζήτημα και δέχομαι ε, τις προτάσεις ε, που έλαβα για την τροπολογία 14. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της κυρίας Λάμπερτ, αυτή η προφορική πρόταση που διατύπωσε δηλαδή, είναι μια πρόταση την οποία μπορώ να δεχθώ, αλλά με τους κατάλληλους τεχνικούς όρους. Για, τις, ε, για την τροπολογίες 15 και 19 βέβαια, θα χρειαστεί ε, να διαβολευτούμε περαιτέρω μεταξύ μας, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να βρούμε συμβιβασμούς. Ολοκληρώνοντας. Λάβαμε 31 τροπολογίες. Δύο εξ αυτών μας δημιουργούν αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Και όταν λέω πρόβλημα εννοώ απλά ότι ε, πρέπει να τη συζητήσουμε ε, περισσότερο αυτές τις τροπολίες, αλλά ε, έχουμε ένα δεκαπενθήμερο μπροστά μας και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, τέλεια. Άρα θα συντάξει τις συμβαστικές προτάσεις, θα τις εξετάσουμε στις 5 Δεκεμβρίου και θα τις ψηφίσουμε αμέσως μετά 16-17 Δεκεμβρίου νομίζω ψηφίζει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στόχος είναι η έκθεση να είναι στην Ολομέλεια τον προσεχή Ιανουάριο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Οπότε περνάμε στο σημείο 24, ε, συγγνώμη, όπου εξετάζουμε το σχέδιο νομοδότησης ε, της ε, Επιτροπής μας για μέκτηση ιδίας πρωτοβουλίας Επιτροπής ΙΤΡΕ με θέμα σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλιβουργία στην Ευρώπη συντάκτη τη γνωμοδότηση εκ μέρου τη Επιτροπή μα είναι ο Πατρίκ Λεϊαρίκ, ο οποίο και θα μας παρουσιάσει τις έξι συμβιβαστικέ προτάσει, ε, οι οποίες προέκυψαν ε, από τι 77 τροπολίε που είχαν κατατεθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους και όσους από εμάς ε, συμμετείχαν στο να εμπλουτίσουμε με τροπολογίες αυτήν την έκθεση. Όπως είπατε, 77 τροπολογίες που βλήθηκαν για ορισμένες από αυτές ε, ταυτίζονται οι απόψεις μας για ένα ή δύο ζητήματα έχουμε διαφορετικές απόψεις θα ξεκινήσω από τα σημεία σύμπτωση. υπάρχει συνένεση για το αιτίε των δυσκολιών λόγω της ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης ε, ο ανταγωνισμός ε, μεταξύ παραγωγών χωρών, ε, τρίτων χωρών που παράγουν χωρίς τα ίδια κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι περιορισμοί στο θέμα των εξαγωγών των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την παραγωγή χάλιβα, και επίσης σημειώνουμε και τις ελλείψεις επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη συμφωνούμε ότι αυτή τη στιγμή σε, είμαστε εισαγωγής χάλιβα δεν υπάρχει λόγος να μειωθεί η παραγωγή μας Αυτά τα δικαιώματα λοιπόν διατήρησης και μάλιστα αύξηση της ε, τρέχουσας ικανότητας ε, έχουμε συμφωνήσει για την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη και για την επιδίωξη εξέβρεσης νέων υλικών για τις ε, πραγματικές διαδικασίες, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Μια δεύτερη σειρά παρατηρήσεων όλοι συμφωνούν ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες για το Χάλεβα ε, βάσει του σχεδίου που προτείνει η Κομισιόν για το Χάλεβα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν για αυτό το σκοπό όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Τρίτη σειρά ερωτημάτων και εκεί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συνένεση. Το πρόβλημα αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις και εντός της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητείται πολύ το θέμα αυτών των κρατικών ενισχύσεων. Είχαμε πει την τελευταία φορά ότι σε ορισμένε παραγωγές όπως το αλουμίνιο συνεχίζουν οι κρατικές ενισχύσεις ενώ ουσιαστικά για το χάλιβα απαγορεύονται. Ορισμένοι από εμάς λοιπόν θεωρούν ότι αν επιτρέπονταν κρέτικες ενισχύσεις για το Χάλιβ διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισμός και ότι κάτι τέτοιο θα άλλαζε το κόστος. Εγώ παραμένω πιστό στην ιδέα ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα με καθαρό πνεύμα μεγάλες χώρες σήμερα συνεχίζουν να βοηθούν τη βιομηχανία της παραγωγή και την χαλιβουργία. Επίσης ε, δεν ε, καταλαβαίνουμε πως κατέχει θα βοηθούσε στο να ενισχύονται ορισμένοι τομείς και όχι άλλοι. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας συνέβαλε θετικά δεδομένου του σημερινού περιβάλλοντος ε, αν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για αυτή την πρόταση η οποία μάλιστα πρέπει να πω ότι συμμορφώνεται με ένα ψήφισμα ε, που είχαμε υιοθετήσει στην Ολομέλεια στις 13 Δεκεμβρίου του 2012 Εκείνη την εποχή λοιπόν έτσι ζητήθηκε να επανεξεταστεί η χαλιβουργία ώστε το μέσο μπορούσε να λαμβάνει κρατικές ενίσχυσεις. Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτό. Το τελευταίο σημείο αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Τον συμπεριλάβαμε ώστε να τονίσουμε το πνεύμα της γνωμοδότησης που ψηφίσαμε μαζί του Αλεσάνδρου Σέρκας Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο πνεύμα και σε αυτό εδώ το κείμενο. Στην πρώτη εκδοχή λοιπόν ε, στην πρώτη εκδοχή των συμβιβασμών λαμβάνουμε υπόψη όλες τις προτάσεις που έγιναν, που εμπλουτίζουν το κείμενο, επιτρέπουν τη συζήτηση τώρα για τα σημεία όπου συμφωνούμε λιγότερο. Προτείνω να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό τόπο για το γενικότερο συμφέρον της χαλιβουργίας της απασχόλησης και των μισθωτών τομέα αυτού. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και βάσει τη συζήτηση που είχαμε μπορούμε να κυκλοφορήσουμε νέες ε, προτάσεις και να συνεχίσουμε να ακούμε ένα τον άλλον και να ανταλλάξουμε απόψεις ώστε να βελτιώσουμε το κείμενο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ. Σαρία Σαϊά και Φιλμπένιον. Σαρία Σαϊά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορούμε πιστεύω να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι απαραίτητο ένα σχέδιο δράση για τη χαλιβουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο κύριος συζήτητης δεν υπογραμμίζει αυτούς αυτά τα σημαντικά στοιχεία το ότι πρέπει να παράσουμε βοήθεια στη Χαλιβουργία στην έκθεσή του και επίσης αυτές οι τροπολογίες συμβαστικές που έχω μπροστά μου είναι τέτοιες που πραγματικά πρέπει να τις συζητήσουμε διαφορετικά η ομάδα του ΕΛΚ δεν θα μπορέσει να τις στηρίξει θα ήθελα να ξεκινήσω με τη συμβιβαστική Α που ουσιαστικά κατηγορεί τη διοίκηση των ε, βιομηχανιών ε, ότι εστιάζεται στο κέρδος εις βάρος των επενδύσεων και των ε, αμοιβών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Γνωρίζουμε όλοι ότι το κόστος της ενέργειας και ότι οι περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν τεράστιες επιτήσεις για τη χαλιβουργία. δεν έχουν συνοχή οι πολιτικές μας και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον όλα αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τομέα αυτά πρέπει να επισημάνουμε και όχι να κατηγορούμε τη διοίκηση δεν καταλαβαίνω πού βασίζονται αυτές οι κατηγορίες ότι η διοίκηση βασίζεται περισσότερο στο κέρδο, εστιάζεται στο κέντρο ει βάρο των επενδύσεων και των αμοιβών. Οι που προσπαθούν να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον. Η συμβιβαστική Β τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι τόσο πολύπλοκη που δεν καταλαβαίνει κανείς σε τι αποσκοπεί αυτή η συμβαστική βήτα. Και εδώ εκτοξεύονται κατηγορίες. Πρέπει να δούμε τι θέλουμε να επισημάνουμε, αλλά χρειάζεται να διάρθρωση αυτή η συμβαστική. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούμε να πούμε εδώ πέρα με αυτή τη συμβαστική βήτα. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για εκ νέου επενδύσεις και τώρα ο εισηγητής λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ενώ ταυτόχρονα κατηγορούμε τις κρατικές ενισχύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να επαναδιατυπώσουμε την όλη συμβαστική Β. Γιατί η συμβαστική Σ δεν συμφωνεί η ΕΛΚ με την εισαγωγή της επιλογής των ε, δημόσιων εξαγορών. Είναι κάτι που ανοίξει το παρελθόν, δεν μπορώ να υποστηρίξω μια τέτοια πρόταση. Στη συμβαστική D θα χρειαστεί να την εξετάσουμε επίσης. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και για τη συμβαστική D. Μετά υπάρχει συμβαστική ε, ε την οποία μάλλον δεχόμαστε περισσότερο από όλες τις άλλες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος αναφέρεται trading, ενώ θα έπρεπε να είναι training, όχι εμπορία, αλλά εκπαίδευση. Και η τελευταία συμβαστική. Θα ήθελα να μου πείτε από πού προέρχονται τα στατιστικά στοιχεία γιατί έχουμε εδώ μία δήλωση αρκετά ισχυρή όπου λέει ότι οι εργαζόμενοι στις τομέα της Καλλιβουργίας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να απολυθούν, να εκτεθούν σε σωματικούς κινδύνους και να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας. Αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, καλό θα ήταν να τα έχουμε εδώ, ότι σύμφωνα με την τάδε μελέτη έχουμε καταλήξει αυτά τα συμπεράσματα. Αλλιώς ε, μάλλον μοιάζει περισσότερο με άποψη παρά με ε, κάτι βέβαιο. Έχουμε πολλή δουλειά όπως είπε ο κύριος συγητής ε, και ευχαριστώ σας συνεργαστώ και εγώ για την αναδιατύπωση και θα σας δώσω και τις απόψεις μου για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε αλλά υπό την παρούσα μορφή των συμβαστικών δεν μπορώ να τις δεχτώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φιλμπένιον Φεντρίκ Και εγώ επέβαλα διάφορες τροπολογίες για αυτή τη γνωμοδότηση με βάση αυτά που είχα πει όταν συζητήσαμε το σχέδιο γνωμοδότησης ακριβώ. Πρώτον, έχω μια τροπολογία που αναφέρεται σε άλλες δυσχέρειες ε, του χαλιβουργικού τομέα. Ευχαριστώ που έγινε δεκτό. Άρα εδώ επετέχθη πρόοδος. Η κυρία Εσάια επίσης ε, το ανέφερε. Να μην πούμε ότι για όλα αυτά είναι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων. Επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα, τις, τα συνδικάτα και για την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενέργειας και όχι μόνο για την εκπαίδευση. Αλλά ίσως να έχω και άλλα σχόλια βαστική Β. Και άλλα πρέπει να κάνουμε για αυτήν. Τρίτον, για τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες κρατικές ενισχύσεις πριν ζητήσουμε αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν οι κρατικές ενισχύσεις είναι ο σωστός τρόπος για να συμμετέχουν ε, οι εργαζόμενοι στη λήψη αποφάσεων και τα υποπτικά συμβούλια. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία ως έχει για τη συμβαστική δέλτα. Θα προτιμούσαμε να επανέλθουμε σε αυτά που υπήρχαν στην έκθεση πρωτοβουλίας, δηλαδή νομικές πράξεις, όχι νομοθεσία. Συμβαστική ε, η τροπολογία μου 60 νομίζω έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη. Αναφέρεται στις μελλοντικές ανάγκες της χαλιβουργίας. Η συμβαστική ε είναι αρκετά αποδεκτή. Η συμβαστική F. Αυτές οι λέξεις για το πόσο σκληρή και ε, αγχωτική είναι αυτή η εργασία. Το ήδη αγχωτική ε, είναι επαρκές. Η κυρία Εσάια είχε δίκιο όταν είπε ότι ήθελε να δει ποιες είναι οι πηγές μας. Άρα πρέπει να κάνουμε ακόμη αρκετή δουλειά, αλλά ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Ε, Νταρντέν και μετά Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις συμβαστικές προτάσεις και τη συνόψιση των κυρίων σημείων που ανέφερε στις τροπολογίες. μερικά στοιχεία που θα ήθελε να συμπεριληφθούν η σοσιαλιστική ομάδα. Ορισμένα έχουν ήδη συμπεριληφθεί, αλλά όχι. Αλλά να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθούν τα κείμενα. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό να αναφερθούμε στον κοινωνικό διάλογο, στην έκθεση του Αλεχάνδρο Θέρκας. Κάτι άλλο, σημαντικό για μας, χρειάζεται μια πραγματική κοινή βιομηχανική πολιτική, ιδιαίτερα για τη χαλιβουργία με επαρκή πρικοδότηση, συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με κανόνες που θα πρέπει να βοηθήσουν ούτως ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να επιτρέψουν ε, μια νέα όθηση για αυτό το τομέα και κανόνες για τον ανταγωνισμό και τον dumping που διαπιστώνουμε. Να μπορούμε δηλαδή να υπερασπιστούμε τον τομέα. Συνολικά, οι τροπολογίες των συναδέλφων μου πιστεύω ότι είναι αποδεκτές δύο θέματα που δεν εθίγησαν από τον εισηγητή στην παρουσίασή του είναι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Θα ήθελα λοιπόν η Ένωση να υιοθετήσει μια ισορροπημένη θέση. Βεβαίως να είμαστε στην πρώτη γραμμή για το περιβάλλον. Νομίζω ότι είμαστε σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου που έχουν οικονομική ισχύ. Δεν θα πρέπει όμως να μας γίνει έμονη ιδέα σε αυτό το τομέα. Κατά πόσο είναι επαχθής η εργασία σε αυτό το τομέα, με εκπλήσουν κάποιες τροπολογίες, κυρίως 69-70, που μοιάζουν, ε, μοιάζει να αρνούνται να ληφθεί υπόψη αυτό στην ε, πολιτική μας για την ασφάλεια στον τόπο εργασίας και τις συντάξεις. Οι συμβαστικές τροπολογίες τώρα. Γενικά είμαι αρκετά θετικός έναντι αυτών. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, βέβαια μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, να βελτιώσουμε, να διατυπώσουμε. Αλλά γενικά είναι προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν βάση εργασίας. Σαφώς ευχαριστώ. Jean Lambert. Δεν είμαι σκιώδης ε, για το θέμα αυτό. Ο κύριος Κορνέλησεν δεν είναι παρόν. Αλλά διαβάζοντας έχω μια-δυο ερωτήσει για το πεδίο εφαρμογής κάποιων, το εύρος κάποιων από αυτές τις τροπολογίες. Είναι ένα θέμα που θέτει η πολιτική μου ομάδα για ορισμένα θέματα, όπως ξέρετε. Ορισμένες τροπολογίες νομίζω είναι περισσότερο θέματα πολιτικής περιβάλλοντος ή βιομηχανίας. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η εκπαίδευση, η διοίκηση των επιχειρήσεων, η κατάρτιση δηλαδή. Αυτά, κυρίως η κατάρτιση, καλύπτεται καλά. Τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων δεν θα σας εκπλήσει ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται και τι ύψους πρέπει να είναι αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή ποιο, ε, ποιες προτάσεις κάνει για το πεδίο εφαρμογή κάποιων από αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Ίσως απλώς να σας πω ότι στις εργασίες μας ε, τον τελευταίο καιρό όπως για παράδειγμα τροποποιήσαμε την πρόταση της Επιτροπής για την ε, μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση όπου αναφερθήκαμε στο ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να πάρουν στα χέρια τους, να πάρουν την ιδιοκτησία μιας επιχείρησης που αντιμετωπίζει τις χέρες, δεν λέω την εύκολο αυτό σε χαλιβουργία, οι εργαζόμενοι να αγοράσουν μια χαλιβουργία, αλλά είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να αναφερθεί στα πλαίσια αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Αν και βεβαίως δεν είναι ένα θέμα που τονίζει το σχέδιο δράσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά με βάση αυτά που είπαμε και για την έκθεση Θέρκας είναι μια ιδέα, ένα μήνυμα που η Επιτροπή μας θα ήθελε να περάσει. Δεν υπέβαλα βέβαια μια τροπολογία για το θέμα αυτό, αλλά εάν σε κάποιο συμβασμό ή με κάποια προφορική τροπολογία μπορούσαμε να το αναφέρουμε, νομίζω πως θα είχε έννοια. Θέλει να μας πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα γίνεται η πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση για την δευτέρα ομάδα υψηλού επίπεδου και έχουμε από κοινού ε, εκπροσώπηση ε, των επιχειρήσεων και των συνδικάτων ε, θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του σχέδιου δράσης. Δεύτερον, κρατικές ενισχύσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι όπως και η ίδια αναφέρατε στις τροπολογίες, η ίδια αναφέρατε στις Έχουμε συζήτηση για την αδιάθρωση των κρατικών ενισχύσεων. Είπατε και εσείς, είπε και ο εισηγητής, ότι γίνεται έντονη εσωτερική συζήτηση στο εσωτερικό της Κομισιόν και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι διαβουλεύσεις. Άρα, πριν το πρώτο τρίμηνο ή τετράμινο, στου επόμενου δεν θα έχουμε κάτι νεότερο. Βέβαια, γνωρίζετε ότι ο τομέα τη Καλλιβουργία ήδη εποφελείται δύο ειδών κρατικών ενισχύσεων, έρευνα, ανάπτυξη και περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δομές του κοινωνικού διαλόγου, γνωρίζετε ότι πιέζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τον κοινωνικό διάλογο έχει συγκληθεί για τη 12η Δεκεμβρίου συνάντηση και κοινωνικό διάλογο στον τομέα της χαλιβουργίας ε, θα είναι παρόν συντονιστής από την Κομισιόν και εκπρόσωποι συνδικάτων και εργοδοσίας. Ε, με το μόνο με το οποίο διαφωνούμε είναι το γεγονός ότι ε, γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνεί να αναφέρονται οριζόντια ζητήματα όπως η πρόταση νομοθεσίας για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε περίπτωση αναδιάδρασης σε ειδικά ε, τομεακά μέτρα για το σχέδιο δράση για τη χαλιβουργία, ολοκληρώνοντας για την κατάρτιση, ε, κοινωνικές πτυχές στον τομέα της χαλιβουργίας. Θα ήθελα να σας πω ότι το ποιοτικό πλαίσιο ε, για την πρόβλεψη αλλαγών ενόψη αναδιαρθρώσεων είναι στη μερίσια της, στην διάταξη της Κομισιόν για τις 10 Δεκεμβρίου. Έχει υπάρξει μάλιστα και προκήρυξη διαγωνισμού για τις δεξιότητες. 15 Ιανουαρίου κλείνει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, ε, προηγουμένως όμως να απαντήσω σε αυτό που είπε η Κομισιόν για την οριζόντια νομοθεσία, για τις αναδιαρθρώσεις, ότι δεν θα πρέπει να περάσουμε σε τομεακές κλαδικές προσεγγίσεις, ε, αλλά μόνο οριζόντια ε, προσέγγιση. Στην πράξη αυτό δεν είναι ακριβές, διότι έχουμε πολλά παραδείγματα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε την τομεακή, την κλαδική νομοθεσία για να προχωρήσει σε θέματα που θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μιας οδηγίας πλαισίου, όπως δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και όχι μόνο. Δείτε την ενημέρωση των εργαζομένων, τη διαβούλευση με τους εργαζομένους. Μπορεί να είναι οριζόντιο το θέμα, να ήταν αντικείμενο μιας οριζόντιας και μόνο αναφέρας, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι σε διάφορα νομοθετήματα τελικά αυτές τις αρχές ε, τις ε, κατανέμουμε, τις ε, υποδιαιρούμε και τις περιλαμβάνουμε στις διάφορες, στις διάφορες νομοθεσίες. Πράγματι, επίσης, όπως είπε η Τζιν Λάμπερτ, ε, υπάρχουν πολλές τροπολογίες, 12 συγκεκριμένα, από την κυρία Σάια και από τον κύριο Νταρντά, θα πρέπει να κρυθούν μη παραδεκτές αφού προηγήθηκε ένας ενδελεχής έλεγχος της γραμματείας και η Προεδρία της Επιτροπής μας επικύρωσε το συμπέρασμά τους. Εκτός βέβαια αν γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε χρόνο και χρήμα ε, για να γίνουν συμβατές, αν δεν γίνει αυτό θεωρούνται μη παραδεκτές. Ο εισηγητής έχει το λόγο, ε, λέει η Αρίκ. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και για τις προτάσεις τους. Δεν έχουμε συμβαστικές τροπολογίες ε, που να έχουν παγιωθεί, αν θέλετε, προς το παρόν τουλάχιστον. Έχουμε μια σύνθεση ε, των τροπολογιών που είχαν κατατεθεί, τις οποίες και λάβαμε υπόψη ώστε να καταλήξουμε στους καλύτερους δυνατούς συμβιβασμούς. Έχω τώρα δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρόκειται περί γνωμοδότησης. Εμείς μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν απαγορεύεται η Επιτροπή μας να εκφράσει την άποψή της. Ανεξαρτήτως του τι θα ε, γνωμοδοτήσουν άλλες επιτροπές και μετά και η Ολομέλεια. Δεύτερη παρατήρηση. Φυσικά και υπάρχει ένα πρόβλημα παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που εισάγουμε. τώρα βέβαια ε, ακούω αυτό το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η διαφορά ε, στο κοινωνικό περιβαλλοντικό ε, επίπεδο δυσχεραίνει τα πράγματα, αυξάνει κάποια χάσματα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε με τα κοινωνικά κριτήρια και τις κοινωνικέ προδιαγραφέ. Εντάξει, μπορεί κανείς να το υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα μέσα στο υφιστάμενο σύστημα και πλαίσιο. Όμως, δεν νομίζω ότι στη γνωμοδότησή μας δεν μπορούμε να πούμε ότι θα θέλαμε να υπάρχει μια παραγωγή ορθότερη, αφού έχουμε στα, στη διάθεσή μας τα τεχνολογικά μέσα. Στη Γαλλία είχαμε ένα παράδειγμα όπου και η γαλλική κυβέρνηση Νομίζω μάλιστα ότι στήριξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα έργο, ένα σχέδιο ε, για ε, μία μονάδα στο Φλωράνζ, αλλά τελικά από τον εργοδότη ε, να βάγισε η όλη προσπάθεια. Λέτε να μην κατηγορούμε τη διοίκηση. Εγώ ξέρετε είμαι επικεφαλής μιας επιχείρησης. Ξέρω γιατί μιλάω. Όμως, οι ιδιοκτήτες, ναι, οι ιδιοκτήτες έχουν στόχους που δεν είναι πάντοτε υπέρ της διατήρησης της παραγωγής και της αναζήτησης ε, περιθωρίων κέρδους. Μπορούμε να το πούμε, δεν υποχρεωτικό, αλλά είναι ένα δεδομένο. Θα ήμουν υπέρ την πρόταση της Προέδρου να τη συμπεριλάβω σε μια συμβιβαστική πρόταση, την πρόταση της Προέδρου μας κυρίας Περβάς Μπερές, για αυτό που λέμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, αυτό που είπατε για τις επιχειρήσεις, να παίρνουν τα ενία εργαζόμενα. Όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας και τα λοιπά, νομίζω ότι Εν γέννη συμφωνούμε. Λέτε να διεξαχθούν μελέτες ε, για το στρες, ε, για την, ε, τα βαρέκια ανθιγυνά ή τέλος πάντων αυτό το χαρακτηριστικό αυτού του επαγγέλματος. Μπορούμε, μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία και να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Έχουμε πάντως μπροστά μας ακόμη κάποιες ημέρες ώστε πραγματικά να υποβάλουμε συμβιβασμούς ε, με την πλήρη έννοια του όρου. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι έχετε ακόμα μερικές ημέρες διότι θα ψηφίσουμε ε, το σχέδιο γνωμοδότησής σας ε, στις 5 Δεκεμβρίου. Αλλά δεν θα συζητηθούν πλέον οι τροπολογίες. Θα πρέπει να ψηφίσουμε απευθείας. Η Επιτροπή η ψηφίζει 16 Δεκεμβρίου. Ολοκλώσαμε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και δίνω λοιπόν τώρα το λόγο για το σημείο 25 όσον αφορά την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σε σχέση με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Δίνω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτριά μας, Σαρία Σαγιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο τριμερής διάλογος πήγε πολύ καλά, πρέπει να παραδεχτώ. Μάλιστα ήταν και πολύ σύντομος χθες το βράδυ τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το ζήτημα αυτό, το θέμα αυτό είναι πολύ τεχνικό. Συνεπώς δεν έγιναν πολιτικές συζητήσεις ε, μεταξύ ομάδων. Συμφωνήσαμε όλοι και υποστήριξαμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Πολύ καλά πρέπει να πω. Για μας, ε, για το Κοινοβούλιο ήταν πολύ σημαντική η αιτιολογική σκέψη ένα θέλαμε να λέγεται στην αρχή ότι τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας δεν πρέπει να θεωρούνται περιορισμοί, ότι αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να φτύγουμε με όλες τις εξαιρέσεις σε όλες τις αγορές εργασίας ανεξαρτήτως επιχείρησης. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο πολιτική δήλωση που κάναμε. Κατά τα άλλα, οι εργασίες εξελίχθηκαν πολύ ομαλά και ικανοποιητικά για Πιστεύω ότι όσοι χρησιμοποιήσουν αυτή την νομοθεσία θα διαπιστώσουν ε, πόσο πιο πρακτική είναι. Κορεπέρ ε, θα λάβει χώρα στις 4. Ε, η ψηφοφορία μας δηλαδή θα, θα είναι όχι την επόμενη μέρα αλλά την εβδομάδα μετά το κορεπέρα, αφού θα έχουμε όταν θα έχουμε την επόμενη συνάντηση τη Επίτροπη Απασχόλησης. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν πολύ ικανοποιητικό και μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή, σε αυτή την οδό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, υπάρχουν ερωτήσεις για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Όχι, όπως καταλάβατε λοιπόν, οι διαπραγματεύσει έγιναν στο πλαίσιο τριμερού διαλόγου. Ίσως όσο πιο τεχνικό είναι ένα θέμα, τόσο πιο εύκολο είναι να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και έναν άλλο τριμερή διάλογο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Πρόκειται για τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας προς τους Άπορους. Δίνω το λόγο στην εισηγητριά μας, Έμαρ Κοστέλο, για να μας αναφέρει την έκβαση του τρίτου τριμερούς διαλόγου. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητριά. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως είπατε, έλαβε χώρα ο τρίτος τριμερής διάλογος για το Ταμείο για τους Άπορους την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβουργού. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος. Ε, είναι πολύ φιλόδοξη εργασία. Ευχαριστώ τους κοιόδης, τις ομάδες και όλο το προσωπικό για τη βοήθειά τους. Έγιναν και πολλές τεχνικές συναντήσεις που βοήθησαν ιδιαίτερα να επιταχύνουμε ορισμένες από τις διαδικασίες. Όπως αναφέραμε ήδη, το Συμβουλίο είχε κάνει κάποιες διαφορετικές νέες προτάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα. Η βασική πτυχή ήταν ουσιαστικά η πρόταση για ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για, την κοινωνική, για δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης ιδιαίτερα για χώρες που δεν ήθελαν να διανύμουν ε, ε, διατροφική βοήθεια. Θέλαμε να το δεχτούμε βάσει ότι αυτές οι δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης δεν, πρέπει να, δεν πρόκειται να επικαλύπτονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα στοχεύει συγκεκριμένα και αποκλειστικά τους άπορους. Είμαστε ικανοποιημένοι με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις ε, που προωθούνται εκεί. θα τις υποστηρίξουμε όλες αυτέ τι διασφαλίσεις και τις θεωρούμε ότι αποτελούν καλή λύση. Επίσης, όπως ανέφερα προηγουμένως, ε, έχω αναφέρει παλιότερα, κοιτάμε την ε, αναθεωρημένη δημοσιονομική ε, κατανομή 3,5 δις έχουν προταθεί από το Σύμβουλο και την Επιτροπή και γίνεται δεκτό αυτό, αντί για 2,5. Και οι μεταβατικές διατάξεις επίσης αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση ε, ορισμού το Κοινοβούλιο έκανε κάποιες αλλαγές στην αρχική πρόθεση της Κομισιόν και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έγιναν δεκτές. Ένας από τους ε, κύριους τομείς είναι η έννοια της εταιρικής σχέσης, η μπλοκή ενδιαφερομένων και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να μειωθεί, να υποβαθμιστεί αυτή η έννοια της εταιρικής σχέσης. Επίσης είχαμε την πρόταση σε σχέση με τις δωρεές τροφίμων που διαφορετικά θα περίπτονταν και ανάπτυξη συνεργειών για το σχετικό τομέα και εδώ προσπαθούμε να εκπονήσουμε προτάσεις που θα διασφαλίζουν τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Επίσης εξετάμε τις συνεργασίες ε, με πολιτικές υγιούς διατροφής, ε, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα απαγορευτικοί ή περιοριστικοί προς τους οργανισμούς αποδέκτες, γιατί θέλουμε να είμαστε βεβαίοι ότι οι δικαιούχοι δεν θα φορτωθούμε υπερβολικό διοικητικό άκθος. Θέλουμε να μπορούν να αναπτύξουν συνεργατικές σχέσεις σε αυτούς τους άλλους τομείς. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο και ειδικότερα για το ζήτημα των κατεξιώδης και εκτελεστικών πράξεων προσπαθούμε να επιλύσουμε μια σειρά από τα ζητήματα που ανέκυψαν σε σχέση με τις πράξεις αυτές πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία. Αναμένουμε κάποιε διευκρινήσει όσον αφορά το ζήτημα που συζητήθηκε λεπτομερώς ε, στην τελευταία συνάντησή τη Επιτροπής Απασχόλησης ε, για τα κοινωνικά για τα κοινωνικά προπολία. Ε, αναφέρθηκε στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής ότι θα διερευνήσουμε τον τομέα αυτό και θα προσπαθήσουμε να τον διευκολύνουμε είχαν σοβαρέ αντιρρήσεις για αυτή την ιδέα το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Η Κομισιόν πρόκειται να προετοιμάσει ένα σημείωμα για μα σε σχέση με τα εμπόδια που υπάρχουν για το ζήτημα αυτό. Όπως ανέφερα, ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε τον τελικό τριμερή διάλογο Υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να εξομαλύνουμε, αλλά μα πιέζει ο χρόνο με αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν. Εάν υπάρξουν. Θέλουμε και οι ΜΚΑ όμικρο να ενημερωθούν γιατί θα υπάρξει υποστήριξη για αυτό το συγκεκριμένο ταμείο. Ε, ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσει για αυτόν τον λεπτομερή πλήρη ε, απολογισμό. Κυρία Ισαριά. Ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις. Μία ερώτηση. Γιατί καθυστέρησαν οι διαπραγματεύσεις για τις πολιετής ε, δημοσιονομικές προοπτικές και άρα και για αυτό το νέο ταμείο. Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ε, να υπάρξει καθυστέρηση στην εφαρμογή του νέου προγράμματος, δηλαδή οι τράπεζες τροφίμων να μην μπορέσουν να αρχίσουν να λειτουργούν την 1η Ιανουαρίου, πόσο καιρό μπορεί να καθυστερήσουν. Φυσικά τα κράτη-μέλη φέρουν την ευθύνη για την ε, ταχεία εφαρμογή των αποφάσεων. Αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση και κενό. Η Πρόεδρος. Άλλες ερωτήσεις. η εισηγήτρια. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Προσπαθούμε να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις. Έχει γίνει η πρόταση. Οι δαπάνες να είναι ήδη, να μπορούν να εκτελεστούν ήδη από τον ε, επόμενο μήνα. Τα κράτη-μέλη ήδη εκπονούν τα προγράμματα ανεξάρτητα από το ότι δεν είχε εγκριθεί οριστικά το πρόγραμμα. Είχαν υπόψη τους όμως τα κράτη-μέλη ότι θα ήταν επιλέξιμη χρηματοδότηση του προγράμματος από 1η Δεκεμβρίου. Το ξέρουν και αυτό τα κράτη-μέλη, ίσως να χρειαστούν λοιπόν κάποιες ε, μεταβατικές χρηματοδοτήσεις. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουν να γίνουν όλα αυτά όσο δυνατόν πιο σύντομα, ώστε οι φιλανθρωπικέ οργανώσει να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότηση. Γιατί ήταν ένα θέμα που μα ενδιαφέρε πάρα πολύ. Θέλαμε οπωσδήποτε, και το είπαμε και στου ε, τριμερεί διαλόγου, ότι θέλουμε να υπάρχουν μεταβατικέ ρυθμίσει. Πρόεδρο. Αυτή είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των τριμερών διαλόγου, δια, των τριμερών διαλόγων. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου επέμεινε ιδιαίτερα να υπάρξουν αυτοί οι μεταβατικοί μηχανισμοί Βέβαια αυτό σημαίνει ότι ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη. Γιατί για να ξεκινήσει η επόμενη περίοδος τα κράτη-μέλη έπρεπε να κάνουν και τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία και την ε, προπαρασκευή των συνθηκών εφαρμογής της. Αλλά παρόμοια ήταν η κατάσταση για το σύνολο των νομοθετικών βάσεων. Όπως είπε η συγγήτρια, εγκρίναμε τις αναγκαίες διατάξεις τις μεταβατικές. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, νομίζω ότι έληξαν οι εργασίες μας, η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 5 ε, και 9 Δεκεμβρίου.